Ja, hallo und Καλησπέρα. Ξέρω ότι πολλοί βρίσκονται ακόμα στο δρόμο. Παρ' όλα αυτά, χαιρετώ όσους είναι παρόντες. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μια τριήμερη συνεδρίαση. Αργό το ξεκίνημα. Θα εγκρίνουμε, όπως συνήθως, την ημερήσια διάταξη έχει σταλεί email που λέει ότι το σημείο 5 θα μεταφερθεί μετά το 7. Πριν το 7, μάλλον συγγνώμη, μετά το 7, αλλά ε, πριν το 6. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη με την τροποποίηση αυτή. Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν. Πέραν του ότι έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από εστονικά και λετονικά. Και φτάνουμε έτσι στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων, όπως συνήθως, εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά των συναδριάσεων 6 και 7 Απριλίου, καθώς και 26 με 28 Απριλίου. Και φτάνουμε έτσι στο πολύ σημαντικό σημείο 4, απολογισμό της επίσκεψης της αντιπροσωπείας ΕΝΒΗ σε χώρα που θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ισλανδία. Ο Ρίχαρτ Ζέιπερ ήταν ε, επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας ε, μαζί με τους συναδέλφους. Θα μας πει ο ίδιος τι αποτελέσματα είχαν το αποτέλεσμα και οι άλλε εκρήξει που έγιναν στην Ισλανδία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είπατε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η επίσκεψη της αντιπροσωπείας αυτής. Ε, είναι... Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε λίγες μέρες ε, είχαμε, αποκτήσαμε μια πολύ καλή επισκόπηση των συνθήκων. Ακούσαμε ε, και τις θέσεις των Ισλανδών ε, σχετικά με την καταστροφή που είχε να κάνει με το ηφαίστειο. Τρεις ε, αντιπροσωπεία από το ΕΛΚ συμμετείχαν στην επίσκεψη αυτή. Οι άλλοι είχαν δυσκολίες λόγω του ηφαιστείου. Ο συνάδελφος Περναντές από την Πορτογαλία ήταν παρόν, καθώς και ο συνάδελφος Φράνκο από την Γαλλία. Επίσης, ε, μας ε, υποστήριξαν ε, διερμηνείς στην επίσκεψή μας αυτή. Όσον αφορά το περιεχόμενο, για να καταλάβει κανείς την Ισλανδία θα πρέπει να κοιτάξει και την ιστορία της. Το 1944 έγινε ανεξάρτητη από τη Δανία η Ισλανδία και γι' αυτό παρά την πολιτική ανεξαρτησία τα αποτέλεσματα των τελευταίων ετών ιδιαίτερα η τραπεζική κρίση οδήγησε στην ε, υποβολή αίτησης για προσχώρηση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρσι, ε, την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο αποφασίστηκε να προσχωρήσει η Ισλανδία. Ήδη έχει υιοθετήσει μεγάλο μέρος του κεκτημένου του κοινοτικού κεκτημένου Ισλανδία. Κάποιοι τομείς χρειάζονται ακόμα προσαρμογές. Ε, δεν ε, σας τα λέω τώρα αυτά, δεν διαβάζω το κείμενο της ε, κυρίας Όλη και να με συγχωρέσει η Γενική Γραμματέα, μερικές φορές οι βουλευτές λέμε και δικά μας λόγια. πάση όσον αφορά την ένβη, έχουμε την οδηγία για την χλωρίδα και την πανίδα. Έχουν εκείνοι απαραίτητες προσαρμογές. Υπάρχουν κάποια ε, προβλήματα προσαρμογής ε, στον ε, τομέα της γεωργίας. Η διάβρωση του εδάφους είναι το σημαντικό πρόβλημα εδώ. Για μας τους Ευρωπαίους ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο τομέας της αλληλείας. Ιδιαίτερα στη δεκαετία του 70 υπήρχαν σοβαρές διαμάχες ε, ιδιαίτερα με τη Μεγάλη Βρετανία λόγω της ζώνης των 300 ε, μιλίων. Το θέμα είναι πιο είναι το αποτέλεσμα της ε, προσχώρησης. Ο έλεγχος και η διαφάνεια θα λειτουργούν πολύ καλά. Δεν είμαι ειδικό στον τομέα της αλληλείας, αλλά από αυτά που είδα εκεί πίστηκα. Πιστεύω ότι η δική μας πολιτική αλληλείας βλέπουμε ότι η αλληλεία της ε, Ισλανδίας ε, λειτουργεί χωρίς επιδοτήσεις. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το περιβάλλον, αλλά επαφευτώσει. Ε, επίσης έχουμε το θέμα των, ε, των φαλενών. Οι Ισλανδοί λένε ότι τα είδη που κυνηγούν δεν απειλούνται από εξαφάνιση και ότι ε, θα πρέπει να εξεταστούν ε, πολύ διαφορετικά ε, οι συνθήκες στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο. Είναι άλλα τα προβλήματα δηλαδή της Αυστραλίας. Η Ισλανδία ισχυρίζεται ότι το 80% των αποθεμάτων των ειδών που κυνηγάει υπάρχουν ακόμα. Αυτά όσον αφορά τις φάλαινες. Ε, πάντως νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα καυτά θέματα στι ε, διαπραγματεύσεις ε, προσχώρησης. Η ενέργεια είναι ε, ενδιαφέρον τομέα. Το 10% της ενέργειας προέρχεται το 10% της ε, ε, Ισλανδικής ενέργειας που προέρχεται από βιώσιμες πηγές ενέργειας ε, καταναλώνεται. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον το ότι υπάρχει τέτοιος όγκος ενέργειας που δεν, που δεν αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης. Νομίζω ότι αυτό θα έχει ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές εταιρείε. Θα είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον ε, να δούμε ε, πώς μπορεί να μεταφερθεί η ενέργεια αυτή στην Ευρώπη χωρίς απώλειες. Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, οι Ισλανδοί έχουν βρει έναν τρόπο λειτουργίας που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός από εμά. Όσον αφορά την διάβρωση του εδάφους, είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Η Ισλανδία έχει αποδασωθεί λόγω ε, οικονομικών δραστηριοτήτων. Απέχουν αρκετά οι Ισλανδοί λοιπόν από μια κατάσταση όπου να μπορούν να διατηρήσουν ε, το έδαφος από τη διάβρωση ε, και να έχουν μια καλή γεωργία. ο Τίμο Σούμα που είναι η επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, της Ισλανδίας. Ε, είναι κάποιος με τον οποίο συναντηθήκαμε επίσης με την Υπουργό Περιβάλλοντος, την κυρία Σβάντης Σβάβαρστοτη που μας εξήγησε πώς έχουν τα πράγματα. Επισκεφτήκαμε γεωργούς ε, ένας μας είπε ότι 20.000 τόνους στάχτης είχε ε, απομακρύνει από ε, τις εκτάσεις καλλιέργειας του και ότι μάλλον άλλες τόσες απέμεναν ακόμα εκεί. Είναι λοιπόν σημαντική η καταστροφή από το ηφαίστειο. Υπήρχαν προβλήματα και με τις επτήσεις αυτό σίγουρα ήταν ε, η σοβαρότερη συνέπεια, αλλά ούτε πολιτικά ούτε με άλλο τρόπο μπορεί κανείς ε, να κάνει κάτι για το πρόβλημα αυτό. Όσον αφορά την ε, πολιτική προστασία φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά. Πολλά βασίζονται σε δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, δικτύωση. Το σύστημα προειδοποίησης ε, του κόσμου ε, φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά, ε, δεν υπήρχαν θύματα παρά την σημαντική καταστροφή. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, τον Ρίχαρτ Σέιμπερ, για την παρουσίασή του αυτή. Βλέπουμε πόσο ενθουσιώδης είναι για την Ισλανδία. Το είδαμε αυτό και στην ε, Ολομέλεια, πώς ε, σωστά επιχειρηματολόγησε σχετικά με τη φαλενοθυρία Μας εξήγησε ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη και ότι αυτά που κυνηγούν οι Ισλανδοί δεν ε, απειλούνται από εξαφάνιση. Τα σημειώνουμε αυτά. Και όσον αφορά το περιβάλλον, ακούσαμε ότι Ε, εφαρμόζονται υψηλής ποιότητας πρότυπα. Ε, το ενεργειακό δυναμικό της Ισλανδίας είναι πολύ ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε αν θέλουν να μας ε, εκχωρήσουν μέρος της ενέργειας τους ή αν μπορέσει να υπάρξει κάποια, κάποιο είδους ανταλλαγή. Ε, ανάμεσα στις χώρες δηλαδή που έχουν ε, ενέργεια από βιώσιμες πηγές ενέργειας ε, και τις χώρες που δεν έχουν τόσο φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας. Η αλληλεία είναι σημαντικό θέμα. Η ποσοστώσεις των ευρωπαϊκών ε, χωρών μπορεί να αποτελέσουν ε, αντικείμενο συζήτηση όσον αφορά τη διάβρωση του εδάφους. Βλέπουμε ότι σε περιπτώσεις αποδάσωσης όπου δεν έχει γίνει αναδάσωση. Υπάρχουν προβλήματα όχι μόνο σε τροπικές ε, εκτάσεις, αλλά και σε μια χώρα όπως είναι η Ισλανδία. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν το θέμα, αν θα υπάρξουν ε, προγράμματα αναδάσωσης ή αν είναι ήδη πολύ αργά, αν δηλαδή δεν είναι αρκετά γόνιμο το έδαφος. Όσον αφορά την προστασία του τοπίου, της υπαίθρου, υπάρχουν ε, φυσικά πάρκα, βιότοποι, η βιοπικιλότητα σίγουρα είναι θέμα, ιδιαίτερα όσον αφορά την θαλάσσια βιολογία. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή. Να ρωτήσω τους συναδέρφους. Ο κύριος Νέλχαρτ έχει μια παρατήρηση, παρακαλώ. Όχι απαραίτητα για την ε, παρουσίαση, ευχαριστώ όμως πολύ για αυτήν, διότι είναι πολύ σημαντική. Ε, τώρα που βρισκόμαστε στην προετοιμασία των ε, ε διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Ισλανδία, έχω μια πρακτική ερώτηση οι θέσεις σε, για μια αποστολή όταν δεν καταλαμβάνονται. Μήπως θα είναι δυνατόν στο μέλλον άλλοι που επίσης επιθυμούν, ε, που προέρχονται από ε, την ίδια πολιτική ομάδα. Μήπως μπορούν να συμμετάσχουν τελικά ε, διότι όσο περισσότεροι αποκτήσουν μια εντύπωση, τόσο πιο πολύτιμο είναι αυτό. Όσο περισσότερα μάτια, τόσο καλύτερη εικόνα που θα έχουμε. Μήπως θα μπορούσε να εξετάσουμε, μήπως θα είναι δυνατό αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Ρίχαρντ για την εισήγησή του. Μία ερώτηση θα ήθελα ε, να υποβάλω. Μιλήσατε για την εξής δυνατότητα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγονται στην Ισλανδία να μπορέσουν να αποσταλούν κι αλλού. Μιλώ για τη γεωθερμική ενέργεια στην Ευρώπη. Ποιες τεχνολογίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτή τη μεταφορά ενέργειας. Η κυρία Μαρίνα Γιανακουδάκη. Um, Ευχαριστώ. Με ενδιαφέρει πολύ η Ισλανδία. Προέρχομαι από εκλογική περιφέρεια που υπέφερε από την τραπεζική κρίση 27 εκατομμύρια ε, διακυβεύθηκαν. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι πηγαίνει καλά η Ισλανδία όσον αφορά το ηφαίστειο. Ξέρω ότι αυτό που εξεράγει ήταν το μικρό και ότι υπάρχει ένα μεγάλο ε, ηφαίστειο. Ε, τι γίνεται με τις, την έγκαιρη προειδοποίηση, υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο αν πάνε στραβά τα πράγματα, πώ επηρεάζουν αυτά την οικονομία. Και επίση αναφέρατε τον ε, γεωργό με τη στάχτη. Ε, μπορεί κανεί να χρησιμοποιήσει τη στάχτη αυτή, έχει καμιά αξία, μπορεί για παράδειγμα να ναι, ναι, ναι, να μπει στο έδαφος για να το κάνει πιο γόνιμο ή να χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή δρόμων. Ο επικεφαλής αντιπροσωπείας, ο Ρίχαρτ Ζήπερ, θα απαντήσει. Ε, όσον αφορά το θέμα των θέσεων, υπάρχουν οι ποσοστώσεις. Ε, νομίζω ότι η Γραμματεία θα πρέπει να το ε, λύσει αυτό το θέμα, διότι ε, φυσικά κάθε πολιτική ομάδα ε, έχει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων. Ε, δεν ξέρω αν μπορεί να αναλάβει άλλη πολιτική ομάδα τις θέσεις αυτές, αλλά ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε. Εάν άλλες πολιτικές ομάδες θέλουν να χωρίσουν τις θέσεις τους, τότε φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Όσον αφορά την ενέργεια, την ερώτηση του του Βιτόριο Πρόντι. Μιλάμε για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτό οδηγεί σε απώλεια. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, στην πράξη ήδη γίνονται προσπάθειες μεταφοράς της ενέργειας με μικρές απώλειες. Και η Γερμανία εξετάζει σε συνεργασία με Γερμανούς εταίρους πώς ε, θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να τοποθετηθούν ε, αγωγή μεταφοράς της ενέργειας ε, στο βυθό, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί φτηνά και χωρίς απώλειες η ενέργεια αυτή στην Ευρώπη. Το θέμα της πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη εξαρτάται πολύ από την τεχνολογία των αγωγών. Για παράδειγμα, αν έχουμε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στον Νότο, θα πρέπει να μπορούμε να μεταφέρουμε την ενέργεια αυτή σε μεγάλες αποστάσεις. Αν ε, δεν το καταφέρουμε αυτό, θα έχουμε πρόβλημα με την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει εμείς οι ίδιοι. Το πλεονέκτημα των, ε, ε της γεωθερμίας και της ε, υδροελεκτρικής ενέργεια στην Ισλανδία ε, είναι ότι ε, γενικά υπάρχει σταθερή ε, παραγωγή στην Ισλανδία. Συνάδελφοι, όσον αφορά το μικρό ηφαίστειο, αυτό ήταν το ηφαίστειο που εξεράγει πράγματι. Δεν θα τολμήσω να προφέρω το όνομα, αλλά είναι γεγονός ότι αυτό είναι το μικρό ηφαίστειο αλλά ήταν τόσο επικίνδυνο για τις αερομεταφορές μας, διότι υπήρχε τεράστια ποσότητα στάχτης και μάλιστα μια ε, μορφή στάχτης που παραμένει στον αέρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα σωματίδια είναι πάρα πολύ μικρά και δεν ε, ενώνονται με άλλα σωματίδια για να πέσουν στο έδαφος. Ε, μένουν λοιπόν πολύ, πολύ χρόνο στον αέρα και τα ορούμενα αυτά σωματίδια είχαν τόσες τόσο σημαντικές συνέπειες. Η ίδια η έκρηξη δεν ήταν λοιπόν τόσο μεγάλη για, την Ισλανδ, για τους Ισλανδούς ε, οι συνέπειες ε, για την, ε, τις αερομεταφορές ήταν μικρές διότι το νέφος αυτών των σωματιδίων μεταφέρθηκε νότιο-ανατολικά προς την Ευρώπη. Περιφερειακά σημαντικό ήταν το, οι σημαντικές οι συνέπειες στην ε, γεωργία. Τι μπορεί να κάνει κανείς με τη στάχτη αυτή που πέφτει στο έδαφος. Ε, λίγα πράγματα, διότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γίνεται σκληρό σαν μπετόν και γι' αυτό πρέπει να αφαιρεθεί από το έδαφος ε, με μπουλντόζες. μακροπρόθεσμα. Πράγματι αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως λείπασμα, αλλά διαρκεί πολύ το να απορροφηθεί αυτό από το έδαφος υπομορφή που να μπορεί να ε, ωφελήσει την, ε, τις καλλιέργειες. Το άλλο, το μεγάλο ηφαίστειο, ε, απειλεί ότι θα εκραγεί ε, φαίνεται ότι σύντομα θα γίνει αυτό. Υπάρχει, κάποια, ε, υπάρχει κάποιο μοτίβο όσον αφορά την συχνότητα ε, εκρήξεων. Ε, αλλά οι εκρήξεις του ηφαιστείου αυτού του κάκλα ε, χαρακτηρίζονται από το ότι δεν οδηγούν σε αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια που έχουν σημαντικές συνέπειες για τις αερομεταφορές. Και τα δύο ηφαίστεια αυτά αποτελούν πρόβλημα επειδή βρίσκονται κάτω από παγετώνα ε, που, ε, και έτσι λιώνει, λιώνουν μεγάλες ποσότητες πάγου. Είναι εντυπωσιακή η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά τις εκρήξεις των ηφαιστείων αυτών λιώνουν οι πάγοι, κάτι που οδηγεί σε ε, τεράστιους ε, χυμάρους, το οποίο επηρεάζει όλη την ε, υποδομή, τις γέφυρες, τους δρόμους, τα σπίτια. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα των Ισλανδών. Λιγότερο τους, επηρεάζουν, τους επηρεάζει η φεστιακή στάχτη δηλαδή και οι συνέπειες της για τις αερομεταφορές. Όσον αφορά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ε, έχουν ε, κάποιες γεωλογικές ε, μετρήσεις όπως παντού. Ποιος αποφασίζει όμως πότε το σύστημα προειδοποίησης πρέπει να πάρει μπρος για να ενημερωθούν οι άνθρωποι. Από ό,τι φαίνεται, όσον αφορά το ηφαίστειο αυτό, ένας γεωργός πήρε τηλέφωνο και είπε ότι τώρα θα εκραγεί το ηφαίστειο, διότι οι γεωλόγοι δεν το είχαν διαπιστώσει αυτοί. Ένας γεωργός που κοίταζε έξω από το παράθερό του πήρε τηλέφωνο και είπε ότι αυτή τη στιγμή εκρήγνεται το ηφαίστειο και έτσι κινητοποιήθηκε το σύστημα προειδοποίησης ε, και εκενώθηκε η περιοχή. Η δυσκολία από ό,τι μας είπαν είναι ότι οι σεισμογράφοι οι γεωλόγοι δεν μπορούν ε, να προβλέψουν ε, με τις λεπτομέρειες μιας τέτοιας έκρηξης. Η, παρατήρηση, η απλή παρατήρηση πολύ συχνά έχει καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα, μια σύντομη διάλεξη περί του Ισλανδικού ηφαιστείου και ότι εν τέλει τα μάτια των ανθρώπων αξίζουν περισσότερο από τις μηχανές. Σώθηκε όμως και η πτήση σας από εκεί μέχρι Βρυξέλλες γιατί από εκεί που έρχεστε θέλω να πω μέχρι Βρυξέλλες γιατί η επόμενη έκρηξη φεστιού θα ε, οδηγήσει σε έκκληση στάχτης ή τέφρας με λιγότερο μικρά σωματίδια. Ευχαριστώ και τη γραμματεία. Τώρα, ερχόμαστε στο 7 που λέει κάνοντας το σωστό. Σχετικά δηλαδή με τον σχεδιασμό των περιβαλλοντικών επιθορήσεων. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Τίκενς, μέλος του Συμβουλίου και συμπρόεδρο του Better Regulation Cluster και του Rob Kramers που είναι manager και αυτός του ε, σχεδίου, του project κάνοντας το σωστό. Θα μας κάνουν τη σχετική εισαγωγή για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο μας απασχολεί έντονα. Τέκες, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας προσφέρετε να παρουσιάσουμε το έργο μας. Θα σας πούμε κάπως ευρύτερα τα πράγματα από ό,τι είχαμε ανακοινώσει στην αρχή. Βέβαια πάντοτε μέσα στο περιθώριο του χρόνου που μας έχετε δώσει. Νομίζω ότι σας έχουμε δώσει τα, τις διαφάνειες. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν αυτές τις διαφάνειες στην παρουσίασή μας. Το θέμα μας είναι βελτίωση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και σχετικές βελτιώσεις. Θα αναφερθώ πρώτα στην, θα σας εξηγήσω πρώτα ποια είναι η Impel και το Impel Cluster για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και θα έρθουμε μετά σε δύο σημαντικά έργα που και τα δύο αφορούν στην βελτίωση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων στις χώρες μέλη την Impel Review Initiative, όπου γίνονται δηλαδή επιθεωρήσεις από ισότιμες οργανώσεις άλλων χωρών και επίσης το project κάνοντας το σωστό για τον καλύτερο σχεδιασμό των ε, περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Όπως βλέπετε στο τρίτο στην τρίτη διαφάνεια εμείς έχουμε 32 χώρες μέλη και όχι 34. Είναι οι χώρες μέλη λοιπόν και η Κροατία, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της ε, Μακεδονίας, Τουρκία και Ισλανδία. Η οποία Ισλανδία έγινε μέλος μόλις την εποχή που άρχιζε να εκρήγνεται το ηφαίστειο. Πάντως εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που την έχουμε ως μέλος. Είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός σε αυτές τις 32 χώρες και έχουμε και νομική προσωπικότητα το 2008. Πολύ σύντομα, γενικά η αποστολή του δικτύου μας είναι να οδηγήσουμε σε πιο αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και αυτό με διάφορους τρόπους, με την ανάπτυξη των άριστον πρακτικών με την ανάπτυξη ενός οπλοστασίου ε, μιας εργαλειοθήκης για τα θέματα αυτά, για capacity building, για την ε, εκπαίδευση των επιθεωρητών. Επίσης, κάνουμε και κοινέ ενέργειες, δηλαδή διάφοροι οργανισμοί καταβάλουν κοινή προσπάθεια για να κάνουν κοινέ επιθεωρήσεις. Επίσης, αναπτύσσουμε σχέδια ε, δραστηριότητες μέσα στις χώρες με την συνεργασία ή και για τη συνεργασία των περιβαλλοντικών αρχών. Θέλουμε επίσης να δώσουμε το λεγόμενο feedback στους νομοθέτες σχετικά με την εφαρμοσιμότητα ορισμένων πρωτοβουλειών και διερευνούμε και την δυνατότητα χρήσης νέων μέσων, νομοθετικών μέσων. Είναι η βασική μας δραστηριότητα είναι η εκτέλεση των έργων αυτών, 15 με 20 ανά έτος, και είμαστε ανοιχτοί και σε συνεργασία μη μελών. Άρα κάθε ένας ο οποίος εργάζεται στην πράξη σε ένα περιβαλλοντικό οργανισμό σε κάποια χώρα μέλος μπορεί να συμμετάσχει σε τέτοια project. Πολύ σύντομα τώρα για την οργάνωση του δικτύου μας, όπως είπα πρόσφατα αποκτήσαμε νομική προσωπικότητα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχουμε λοιπόν μια γενική συνέλευση. Στη γενική, μα, γενική μας συνέλευση συμμετέχουν όλες οι περιβαλλοντικές αρχές των χωρών μελών μας και εκεί συνέρχονται για να συζητήσουν τον σχεδιασμό των project. Εκεί έχουμε και παρατηρητές οι οποίοι προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον ΟΟΣΑ και από άλλα περιβαλλοντικά δίκτυα. Έχουμε το εκτελεστικό συμβούλιο το οποίο ασχολείται με την καθημερινή εργασία του συνδέσμου, έχουμε επαγγελματίες, επαγγελματίες συγγνώμη, αλλά πολλή από τη δουλειά γίνεται στα τρία κέντρα, στα τρία clusters, ε, όπως ε, αποκαλούνται στα αγγλικά. Έχουμε προγράμματα εργασιών και η βασική μας δραστηριότητα, όπως είπα, είναι η εκτέλεση των διαφόρων έργων, project. Κάθε τρία χρόνια κάνουμε μια μεγάλη συνδιάσκεψη που την οργανώνουμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξηγήσουμε ε, σε ένα ευρύτερο κοινό το τι ακριβώς κάνουμε. Σημαντικό είναι επίσης να πω ότι έχουμε και ένα μνημόνιο συμφωνίας για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθούμε να συντονίζουμε το έργο μας δηλαδή με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών. Τώρα η διαφάνεια 6. Μέσα στην, ε, στον σύνδεσμό μας έχουμε τα τρία λεγόμενα κλάστερ. Το πρώτο αναφέρεται στην, σε εγκρίσεις, επιθεώρηση και επιβολή. Είναι πολύ ευρύς ο τομέας αυτός, δηλαδή ασχολούμαστε και με την επιθεώρηση και με την έκδοση αδειών για την επιθεώρηση και σε την επιθεώρηση βασιζόμαστε στα ελάχιστα κριτήρια των επιθεωρήσεων που είναι ε, σημαντική αναφορά στο έργο μας σχετικά με τις επιθεωρήσεις. Κάνουμε επίσης και πολλή δουλειά σχετικά με τις χορηγήσεις εγκρίσεων σε σχέση με το IPPC, με τα ύδατα κτλ. Το 2 αναφέρεται σε διαμεθοριακές μεταφορές αποβλήτων. Αυτή η ομάδα κάνει ε, και αναλαμβάνει κοινέ δραστηριότητες επιβολής. Εκεί εκπαιδεύουμε κιόλας επιθεωρητές. Και το τρίτο, η τελευταία ομάδα, ε, ασχολείται με την βελτίωση της νομοθεσίας. και ασχολείται με το να αναφέρει, με το να δίνει feedback ε, στους νομοθέτες. Έχουμε ένα κατάλογο κριτηρίων, ένα checklist για την βελτίωση της νομοθεσίας και πρόσφατα κάναμε τη σχετική εργασία για το IPPC και για το WIG Έρχομαι τώρα στο έργο της πρώτης ομάδας, του πρώτου κλάστερ, για τις ε, εγκρίσεις και επιθεωρήσεις, η οποία πρώτη αυτή ομάδα εργάζεται σχετικά με τις επιθεωρήσεις, αναφερόμενη στην Ευρωπαϊκή Σύσταση για ε, τα ελάχιστα κριτήρια, σύσταση την οποία έχει οθετήσει ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και η οποία βρίσκεται σε φάση αναθεωρήσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΙΜΠΕΛ έχει ένα δίκτυο ε, όσων ασχολούνται στην πράξη με τα θέματα αυτά και οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση της βάσης για την σύσταση αυτή με την υποβολή ορισμένων κριτηρίων τα οποία μετά, τελικά μετά από επεξεργασία κατέληξαν να μπουν στην σύσταση και από τη στιγμή εκείνη μια σειρά project για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών επιθεωρήσεων έγινε. Εξακολουθούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα ε, εξέτασης από ισοδύναμες ή ισότιμες αρχές και έχουμε συντάξει και έγγραφα κατευθύνσεων για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Ένα από τα εγγραφτά αναφέρεται και στον σχεδιασμό των επιθεωρήσεων μέσα στο πλαίσιο του κάνοντας το σωστό. Συμβάλλουμε και στην επανεξέταση της σύστασης, την οποία έχει αναλάβει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένες τροποποίησεις του κειμένου με στόχο να ενισχυθεί. Λίγα λόγια τώρα για την πρωτοβουλία επανεξέτασης της ΙΜΠΕΛ, η οποία είναι εθελούσια και έχει ως στόχο να εφαρμόσει ορισμένες διατάξεις μέσα στην ίδια την σύσταση που λέει ότι οι χώρες μέλη προσφέρουν διοικητική αρρωγή για την ε, ε, εφαρμογή της συστάσεως σε σχέση με επιθεωρήσεις με διαδικασίες επιθεωρήσεων που θα βελτιώσουν στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την κοινότητα. Πρόκειται για παροχή συμβουλών δηλαδή, οι οποίες ενισχύουν το έργο των επιθεωρήσεων. Τα πλονεκτήματα τώρα από την Impel Review Initiative, η επανεξέταση αυτή προσφέρει χρήσιμες συμβουλές από αυτούς που ασχολούνται στην πράξη για τις ε, δομές. Μία αρχή μπορεί να επιλέξει την ε, συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο τύπο επιθεώρησης που επιθυμεί, αναλόγως με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται και μπορεί επομένως να αναζητήσει συμβουλές από άλλους αρμόδιους σε άλλες χώρες. Η αναθεώρηση αυτή τονίζει επίσης τις καλύτερες πρακτικές, περιλαμβάνει έναν αριθμό συστάσεων που μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση της οργάνωσης της ε, συγκεκριμένης δημόσιας αρχής και άλλες δημόσιες αρχές μπορούν να διδαχθούν από αυτές τις συστάσεις και από τις βέλτιστες πρακτικές και να τις εφαρμόσουν στα δικά τους δίκτυα. Η Initiative διεξήχθη ήδη σε έναν αριθμό χωρών. Πέρσι έκανε τέτοια πρωτοβουλία επανεξέτασης η Πορτογαλική αρχή, φέτος η Σλοβενική, επίσης η αρχή στη Ρουμανία, την επόμενη χρονιά είναι η σειρά της Λετωνίας και της, Κροτα... και της Κροατίας. Η πρωτοβουλία Impel Review είναι κάτι που θέλουμε να συνεχίσουμε, προσπαθούμε να την βελτιώσουμε, ώστε να γίνει πιο ελκυστική σε ακόμα περισσότερες δημόσιες αρχές στις χώρες μέλη και νομίζω ότι πετυχαίνουμε στο στόχο μας αυτό, διότι έχουμε τώρα πολλές νέες χώρες οι οποίες ζητούν ε, να συνεργαστούμε στην IRI. Είναι σημαντικό για την συλλογή προφοριών και για την διεξαγωγή συζητήσεων μεταξύ της ομάδας που κάνει την ε, επιθεώρηση αυτή και των δημοσίων αρχών. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο. Ακολουθεί τις κατευθυντήρες γραμμές του κάνοντας το σωστό. Επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφό μου δίπλα μου για να σας πει αυτά περί του κάνοντας το σωστό. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω το κάνοντας το σωστό αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα του ΙΜΠΕΛ, έτσι ώστε να προγραμματίσουμε τους ε, περιβαλλοντικούς ε, ελέγχους. Ε, διεξήχθη από την Ολλανδία μαζί με τη Γερμανία, Σουηδία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ουγγαρία. Θα ήθελα εντάχει να σας μιλήσω για θέματα σχεδιασμού ως προς το σχέδιο κάνοντας το σωστό και μετά να μπω σε λεπτομέρειες. Μέσα στα πλαίσια του κύκλου ελέγχου και εποπτείας του περιβάλλοντος. Το τελευταίο τμήμα της παρουσίασης αφορά τη διάρθρωση αυτού του ε, οδηγού ακολουθήσαμε αυτή την προσέγγιση, αυτή την καταβήμα προσέγγιση, διότι αυτό που έχει σημασία είναι η διάρθρωση και τα καθήκοντα των ε, αρχών επιθεώρησης στα κράτη-μέλη γι' αυτό και ο οδηγός είναι ευέλικτος και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Αυτός ο οδηγός, ο βαθμιαίος οδηγός, οδηγεί στο να μπορούν τα κράτη-μέλη να τηρούν τα ελάχιστα κριτήρια προδιαγραφών εποπτείας. επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τα βασικά θέματα προγραμματισμού. Γνωρίζουμε ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι και υπάρχουν, υπάρχει πληθώρα καθηκόντων και ευθυνών. Ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει το input να είναι αποτελεσματικό. Γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε προτεραιότητες. Μετά από αυτό θα πρέπει να ε, δούμε ποιες είναι οι στοχοθετήσεις μας και πώς μπορούμε να τις επιτύχουμε. Όλα αυτά εντάσσονται στο σχέδιο επιθεώρησης. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε πώς προωθείται αυτό το πρόγραμμα, το οποίο άρχισε το 2006 και πέρσι του εδόθη τελική μορφή. Το 2006 ε, αναζητήσαμε τις προτεραιότητες των κρατών μελών σε αυτό το θέμα, της ιεράρχησης δηλαδή προτεραιοτήτων, είδαμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι χρειάζονται κατευθυντήριες γραμμές και το 2007 καταρτήσαμε αυτό τον οδηγό βαθμίας προσέγγισης. Αυτό χρειάστηκε δύο με τρία χρόνια. Αρχίσαμε με ένα workshop εμπειρογνωμόνων. Δείξαμε αυτό τον οδηγό στους εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη και τους ζητήσαμε να προωθήσουν αυτό το σχέδιο σύμφωνα με τη μεθοδολογία τους και να προβούν σε συστάσεις βελτίωσης. Άρα βελτιώσαμε τον οδηγό αυτό και άρχισαν, άρχισε η κατάρτιση από τους άμεσα ενδιαφερόμενους από τα κράτη-μέλη. Ε, οργανώθηκε μια κατάρτιση τριών ημερών. Το 2009 ήταν το έτος εφαρμογής, όπου είχαμε workshops υποστηρίζοντας τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας. Όπως είπε και ο συνάδελφος, προωθήσαμε και την μεθοδολογία του κάνοντας το σωστό. Τώρα στην ιστοσελίδα του Impel προβήκαμε σε ανταλλαγή καλών πρακτικών που ήδη προϋπάρχουν. Ως προς τον κύκλο επιθεώρησης, τον περιβαλλοντικό κύκλο επιθεώρησης, στην διαφάνεια υπαριθμό 15, προέρχεται από τις συστάσεις. Στις ίδιες τις συστάσεις ε, βλέπετε ε, αυτή την, αυτό τον κύκλο του προγραμματισμού, της εκτέλεσης του πλαισίου, της εκτέλεσης και καθοδήγησης, καθώς και της απόδοσης, της εποπτείας της απόδοσης. Το πρώτο κουτί αφορά τον προγραμματισμό. Τι είναι το πιο σημαντικό και τι θέλουμε να επιτύχουμε. Και πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Το επόμενο κουτί αφορά το πλαίσιο εκτέλεσης, δηλαδή τους όρους ε, για τους ε, επιθεωρητές, κατάρτιση, εκπαίδευση, επαρκής εξοπλισμός και ούτω καθεξής. Ως προς την εκτέλεση και την έκθεση δεδομένων, πρόκειται για επιτόπιες επισκέψεις και κατάρτιση εκθέσεων. Ως προς την εποπτεία της ε, αποτελεσματικότητας ή της απόδοσης, μας ενδιαφέρει ποια είναι η έκβαση όλης αυτής της διαδικασίας επιθεώρησης και πώς μπορούμε να εντάξουμε αυτά τα δεδομένα στον οδηγό επιθεώρησης. Αυτός ο κύκλος επιθεώρησης μας δείχνει ότι ο κύκλος του προγραμματισμού ήταν λίγο πιο περίπλοκος και μέσα στα πλαίσια αυτού του κουτιού προγραμματισμού ορίσαμε έναν άλλο κύκλο που βλέπετε στη διαφάνεια 16. Αφορά το έργο της επιθεώρησης, της ευθύνες, της αρμοδιότητες, τον καθορισμό προτεραιοτήτων πώς μπορούμε να επιτύχουμε τους συγκεκριμένους στόχους. Αυτό το βλέπουμε στο 1C. Και αυτό εντάσσεται στο σχέδιο επιθεώρησης γενικότερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο κύκλος προγραμματισμού, ο περιβαλλοντικός κύκλος προγραμματισμού που αφορά τη διαφάνεια υπαριθμό 17. Θα δούμε τα διάφορα στοιχεία Ένα α Πλαισίωση. Ο επιθεωρητής και η αρχή επιθεώρησης θα πρέπει να ορίσει τις αρμοδιότητες και την αποστολή, καθώς και τους στόχους σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να περιγράψουν τον γεωγραφικό τόπο για τον οποίο είναι υπεύθυνοι. Επίσης, θα πρέπει να συλλέξουν πληροφορίες για την κατάσταση του περιβάλλοντος και τη συμμόρφωση ανάλογα με το, τα εφόδια που έχουν στην περιφέρεια αυτή. Όλα αυτά είναι τα στοιχεία εισρωής, το input. Επίσης χρειάζεται μία αποτίμηση κινδύνων που εντάσσεται στην ε, στο άρθρο 23 της αρχικής οδηγίας. Υπάρχει εκεί μια παράγραφος για τις επιθεωρήσεις η οποία ασχολείται με αυτό το θέμα της προσέγγισης ανάλογα με την αποτίμηση κινδύνων, αξιολόγηση κινδύνων στη συχνότητα επιθεωρήσεων. Άρα χρειάζεται αυτή η εκτίμηση κινδύνων και το output μπορεί να ακολουθήσει μία ιεράρχηση, βλέποντας ποιοι είναι και οι διατηθέμενοι πόροι. Το 1C ορίζει τους στόχους και τις στρατηγικές. Όταν ξέρουμε τι είναι σημαντικό, θα πρέπει να ορίσουμε τι είναι το, ποιο είναι, ποιος είναι ο στόχος. Αυτό γίνεται με τις στοχοθετήσεις που έχουμε ορίσει. Αν ξέρουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το επιτύχουμε, έτσι ώστε η προσέγγιση μας να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτική. Αυτό δεν φορά μόνο επιτόπιες επισκέψεις. Θα πρέπει να προωθήσουμε το θέμα της ε, συμμόρφωσης και της επικοινωνίας. Το τελευταίο κουτί, το 1D, είναι εκεί που συμπλέουν τα πάντα όταν υπάρχει δηλαδή το σχέδιο επιθεώρησης, το οποίο δημοσιοποιείται, καθώς και τα επιμέρους προγράμματα επιθεώρησης. Επίσης, η αναθεώρηση είναι απολύτως απαραίτητη, διότι χρειάζεται μία ενημέρωση για να δούμε κατά πόσο τα στοιχεία είναι επικαιροποιημένα και το κατά πόσο δηλαδή έχουμε επιτύχει τους αρχικούς στόχους ή κατά πόσο χρειάζεται μία μερική αναθεώρηση. Η τελευταία διαφάνεια αφορά τον ίδιο τον οδηγό. Εδώ βλέπετε πώς το... ο οδηγός βαθμίας προσέγγισης ορίζεται από τρία βασικά κεφάλαια. Το κεφάλαιο 2 σας δίνει τα, τις πληροφορίες και τις συστάσεις. Στο κεφάλαιο 3 προσπαθούμε να ορίσουμε, να το συνδέσουμε αυτό με τον κύκλο επιθεώρησης που έχουμε αναπτύξει και το κεφάλαιο υπαριθμών 4 οδηγείται στις λεπτομέρειες του, των στόχων της αναθεώρησης και της ενημέρωσης. Όσο πιο λεπτομεριακά διαβάζετε αυτό τον οδηγό, όλα τόσο περισσότερα στοιχεία θα βρείτε. Οι πληροφορίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Ιμπελ. Είναι μια νέα ιστοσελίδα, εργαζόμαστε πολύ σκληρά και ο οδηγός θα είναι διαθέσιμος και στον ιστότοπό μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Ο κύριος Λοπάτα θα ήθελε να παρέμβει τώρα ή αργότερα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα, αλλά πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα κάνοντας το σωστό της Επιτροπής είναι ένα από τα πιο χρήσιμα οικολογικά προγράμματα που εφαρμόζονται, διότι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση ε, των ε, περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Και πιστεύω ότι οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις θα πρέπει όχι μόνο να εκτελούνται, αλλά να ελέγχονται και να γίνονται πιο αποτελεσματικές. Το κάνοντας το σωστό, τα προγράμματα κάνοντας το σωστό, και η ε, ανακοίνωση με τις συστάσεις για περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Τα δύο αυτά συνδέονται στενά. Το δεύτερο αυτή τη στιγμή αναθεωρείται και γι' αυτό η Επιτροπή είναι σε στενή επαφή με την ΙΜΠΕΛ για να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των ε, προγραμμάτων αυτών ε, που θα χρησιμεύσουν ε, κατά την αναθεώρηση των συστάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ποιος άλλος θα ήθελε το λόγο. Ο κύριος Πέτερλε ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Με χαρά άκουσα την παρουσίαση αυτή. Και έχω την αντίποση ότι πράγματι κάνει το σωστό η οργάνωση αυτή. Αυτό που θα ήθελα να ξέρω είναι από τις γνώσεις που προσφέρετε, ποιες είναι πιο χρήσιμες και σε ποιον τομέα πιστεύετε ότι χρειάζεται περισσότερο βοήθεια, ποια είναι τα προβλήματα που είναι πιο δύσκολα να αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι ομιλητές, άλλες ερωτήσεις. Δεν νομίζω. Θα ήθελα και εγώ να υποβάλω μια ερώτηση πριν απαντήσετε. Πέρυσι έγινε λόγος για δημιουργία μιας ομάδας κρούσης στις 8 Οκτωβρίου για τις επιθεωρήσεις και από την άλλη να υπάρχει μία οδηγία ως προς τις επιθεωρήσεις στον τομέα του περιβάλλοντος. Θα ήθελα να ξέρω πού βρισκόμαστε. Και επειδή υπάρχουν ε, σημαντικές ανεπάρκειες στην εφαρμογή του κανονισμού, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο ε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει μία μνήα προς την Επιτροπή, μία έκκληση προς την Επιτροπή έτσι ώστε να συμμορφωθούν οι χώρες που δεν τηρούν τον ε, κανονισμό. Ο κύριος Ζέμπερ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Οι γνώσεις που αποκτώνται από αυτό το δίκτυο πώς εισραίουν στη δουλειά της Κομισιόν. Πώς λαμβάνονται υπόψη, πώς εξετάζονται οι προτάσεις ποιες τροποποιήσεις μπορούμε να διαπιστώσουμε σε σχέση με την κατάσταση πριν την ε, πρωτοβουλία αυτή της questions Οι ερωτήσεις απευθύνονται και στους δύο παρεμβαίνοντες. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στην Επιτροπή και μετά στους συζητητές του σχεδίου. Ο κύριος Λοπάτα, για να, ερω... για να απαντήσει στην ερώτηση του κυρίου Ζέμπερ και στη δική μου. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2007, διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η αναθεώρηση. Η Κομισιόν κάνει μελέτη επιπτώσεων σχετικά με τις διάφορες λύσεις. Εξετάζουμε λοιπόν όχι μόνο την τροποποίηση των υπαρχουσών συστάσεων, εξετάζονται και άλλες λύσεις. που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με την ε, μεταφορά των συστάσεων σε οριζόντια οδηγία ή θα μπορούσαμε να έχουμε σύσταση που να συμπληρώνεται από συγκεκριμένες τομεακές απαιτήσει για τις επιθεωρήσεις με στόχο τους συγκεκριμένους τομούς, το, τομείς που έχουν ανάγκη από νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις. Εξετάζουμε λοιπόν τις λύσεις αυτές, εξετάζουμε και το ευρύτερο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστά. Περιμένουμε η εξωτερική μελέτη αντικτύπου που έχουμε αναθέσει για να πραγματοποιηθεί να ολοκληρωθεί στο τέλος του καλοκαιριού, γύρω στο Σεπτέμβρη. Και η μελέτη επιπτώσεών μας θα είναι και αυτή έτοιμη φέτος το φθινόπωρο. Ανάλογα με τις εξελίξεις, περιμένουμε η πρότασή μας να υποβληθεί αρχές του επόμενου έτους. Φυσικά λαμβάνουμε υπόψη μας, λάβαμε υπόψη μας και λαμβάνουμε ακόμα υπόψη μας τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Περσινές. Αυτή τη στιγμή είναι νωρίς να προδικάσουμε το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Merci. κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως προς το ερώτημα ποιες χώρες χρειάζονται περισσότερη βοήθεια εξαρτάται από το θέμα. Αλλά γενικά όταν πρόκειται για βελτίωση της επιθεώρησης με βάση τις εθνικές αρχές επιθεώρησης ως προς το θέμα, θέματα περιβάλλοντος, οι νέες χώρες χρησιμοποιούν την ε, πείρα των παλαιότερων κρατών μέσω του προγράμματος IRI ή κάνοντας το σωστό. Επίσης, τα νέα κράτη-μέλη ε, ακολουθούν τα δεδομένα που υπάρχουν, διότι ε, κάναμε μία έρευνα IPPC σε σχέση με τις εκμεταλλεύσεις εκτροφής χείρων και είδαμε ότι υπήρχαν διαφορετικές πρακτικές τις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο καθένας και να μάθει από αυτές. Όλα αυτά εντάσσονται στην ε, πολιτική του προγράμματος και οι υπάλληλοι της Κομισιόν συνεργάζονται με τους επιθεωρητές με τους επαγγελματίες του κλάδου έτσι ώστε να ενταχθούν όλα αυτά τα στοιχεία στη γενικότερη διαμόρφωση της πολιτικής. Ως προς τις συστάσεις όπως σας είπα, με βάση την πείρα μας, με την παρούσα σύσταση, έχουμε προβεί προς ε, υποδείξεις για το πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε τη σύσταση, γιατί έμπρακτα ορισμένα στοιχεία δεν είναι απόλυτα σαφή. Άρα προβήκαμε προς ε, συστάσεις που ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη. Και επίσης θέλουμε μία συνεκτική προσέγγιση σε σχέση με τις επιθεωρήσεις, διότι υπάρχουν μεν συστάσεις, αλλά θα θέλαμε στους οδηγούς και στον κανονισμό να λάβουν να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι οι συστάσεις έχουν ενσωματωθεί, είναι ενσωματωμένες. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται κατά ενιαίο συνεπή τρόπο, έτσι ώστε οι αρχές επιθεώρησης στα κράτη-μέλη πρέπει να ε, εφαρμόσουν τους διάφορους κανονισμούς και οδηγίες, να χρησιμοποιήσουν ένα ενιαίο πρότυπο, το οποίο να αφορά όλες τις νομοθεσίες. Και νομίζουμε ότι η σύσταση ή η μελλοντική οδηγία επιθεωρήσεων θα επιτελέσει ακριβώς αυτό το έργο. Δηλαδή να οδηγήσει σε μία συνεκτική ενιαία προσέγγιση ως προς το θέμα των επιθεωρήσεων. Ο κύριος Ζέμπερ. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Ε, κάτι δεν κατάλαβα, ίσως θα μπορούσε να το επαναλάβει ο μιλητής. Από ό,τι καταλαβαίνω το πρόγραμμα αυτό ε, δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επιθεώρηση, έχει να κάνει γενικά με την καλύτερη νομοθεσία. Η Κομισιόν πώς φροντίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού να εισρεύσουν στο, στην νομοθετική δουλειά. Θέλουμε τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας Ιμπερ να οδηγήσουν σε καλύτερη ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε, καλύτερη, σε καλύτερο έλεγχο, καλύτερη εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Euh, Κύριε Λοπάτα, μπορείτε να μας απαντήσετε. Ναι, ευχαρίστως. Το πρόγραμμα Impel κάνοντας το σωστό, εφαρμόζεται στα πλαίσια της δέσμης 1 που έχει να κάνει με την, εφαρμογή των, με την εκτέλεση των ελέγχων, των επιθεωρήσεων. Και δεν έχει άμεσα να κάνει με τη δέσμη 3, την καλύτερη νομοθεσία. Τα αποτελέσματα της δουλειάς της Ίμπελ εδώ και πέντε χρόνια των προγραμμάτων αυτών των τελευταίων πέντε ετών εξετάζονται προσεκτικά στα πλαίσια εκπόνησης των συστάσεων. Και στο πλαίσιο αυτό έχουμε προγραμματίσει μία ε, πρώτη συνάντηση με τους εκπροσώπους της ΙΜΠΕΛ για να εξετάσουμε τη δυνατότητα βελτίωσης ε, της ε, σύστασης. Η σύσταση αυτή δεν αφορά αποκλειστικά τον τομέα του, ε, του προγράμματος κάνοντας το σωστό, αλλά επηρεάζεται από αυτόν. Την επόμενη, τις επόμενες λοιπόν, θα είναι αποτέλεσμα μιας συνάντησης ανάμεσα στην Κομισιόν και τους προσώπους της ΣΥΜΠΕΛ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Άρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους Τίκενς και Κράμερ καθώς και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για αυτή την ε, άκρος ενδιαφέρουσα συζήτηση που δείχνει πόσο αποδοτικοί είμαστε. Περνάμε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης που είναι μία προφορική ερώτηση από τους Evans, McAven και Horst, Schnellhardt, σχετικά με τις επιθεωρήσεις στον τομέα του κρέατος. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή σε πρώτη φάση. Ο κύριος Πουντελέ δεν ξέρω κατά πόσο είναι παρόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν, απαντώντας προς τους τρεις συναδέλφους που υπέβαλαν αυτή την προφορική ερώτηση, θα ήθελα να πω ότι η έκθεση της Επιτροπής του Ιουλίου 2009 είναι μία ε, έκθεση με πραγματικά περιστατικά σε σχέση με το πακέτο περί και υγιεινής και ιδιαίτερα ως προς την διατροφική αλυσίδα και τι επιθεωρήσεις στα σφαγεία. Πρόκειται για μια έκθεση που δεν είναι νομοθετικού περιεχομένου, δεν αλλάζει την παρούσα νομοθεσία ή τον κανονισμό και δεν προβάλλει ε, αντιθέσεις ή τροποποίησεις. Για να απαντήσω, θα ήθελα να απαντήσω στην καθεμία από τις ερωτήσεις ξεχωριστά. Το πρώτο ερώτημα αφορά τις σχέσεις του ε, Γραφείου Κτηνιατρικών Επιθεωρήσεων σε σχέση με θέματα διατροφικής ασφάλειας. Οι εκθέσεις αυτές είναι δημόσιες και η Επιτροπή γνωρίζει ότι υπάρχουν ελλείψεις από τα κράτη-μέλη σε σχέση με την εφαρμογή αυτού του κοινοτικού πλαισίου. Όμως, ο περιορισμένος προϋπολογισμός που ασχολείται με αυτά τα θέματα και η ανεπάρκεια προσωπικού στα κράτη-μέλη δεν εξηγεί αφεαυτού της ανεπάρκειας. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί εδώ και 18 μήνες. Τα κράτη-μέλη θέλουν να μειώσουν το προσωπικό εξαιτίας της ε, οικονομικής κρίσης και Όλες οι διοικήσεις, οι κυβερνήσεις έχουν την τάση μείωσης του προσωπικού. Γνωρίζετε ότι σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επέβαλαν αυτό στις αρχές επιθεώρησης, αλλά υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις αυτού του φαινομένου. Δηλαδή κατάρτιση των επιθεωρητών που είναι ελλειπείς και ούτω καθεξής. Γι' αυτό υπάρχουν αποκλίνουσες εφαρμογές από τα κράτη-μέλη. Όμως είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που μας ανησυχεί και μας ενδιαφέρει η ενιαία εφαρμογή αυτού του πλαισίου, είτε πρόκειται για παλαιά είτε για νέα κράτη, δηλαδή ενιαία εφαρμογή από τους 27 της κοινοτικής νομοθεσίας σε σχέση με την διατροφική ασφάλεια. Αυτή είναι μια κοινή μας ανησυχία, κοινό μας μέλημα και εξαιτίας αυτού του γραφείου κτηνιατρικών αρχών και επιθεωρήσεων έχουμε ε, μία φωτογράφηση της κατάστασης για να δούμε τι πρέπει να διορθωθεί. Ως προς τον, την ανεξάρτητη αυτή αρχή της ε, επιθεώρησης, εμείς συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη, δηλαδή οι επιθεωρήσεις στα σφαγεία θα πρέπει να γίνονται από μία ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει η δυνατότητα για τα σφαγεία που ή κουνελιών να χρησιμοποιήσουν ε, προσωπικό της επιχείρησης μετά από ειδική κατάρτιση, όπως ισχύει και στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων. Και ε, λειτουργούν και δουλεύουν υπό την ε, επιθεώρηση, υπό τον έλεγχο του βασικού επιθεωρητή. Αλλά σε σχέση με τα σφαγεία κόκκινου κρέατος όπως, το, κρέατος όπως το ονομάζουμε, δηλαδή όταν μιλάμε για μοσχάρι, για χοιρινό, για πρόβιο κρέας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το εξής επειδή ακριβώς οι επιθεωρήσεις είναι ελληματικές και επειδή υπάρχει ανεπαρκές προσωπικό, γνωρίζετε ότι η Επιτροπή ζήτησε μία εκτίμηση το 2008, μία αξιολόγηση από μία ανεξάρτητη αρχή των κρατών μελών και αυτά, αυτό το θέμα των ε, τελών επιθεώρησης απασχόλησε τα κράτη-μέλη. Η αξιολόγηση αυτή έδειξε ότι υπάρχει διαφορετική εφαρμογή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρχε δηλαδή εναρμονισμένη προσέγγιση. Γίνεται μία μελέτη αντικτύπου αυτή τη στιγμή για να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει η υπάρχουσα νομοθεσία ε, που λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια, άρα δεν είναι προσαρμοσμένη στις πιο πρόσφατες καταστάσεις και δεδομένα. Θα έχετε και μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου το 2011 και εσείς και το Συμβούλιο. Το τρίτο ερώτημα αφορά αυτούς τους ε, ιδιωτικούς υπαλλήλους ε, σε σχέση με τις επιθεωρήσεις για το κόκκινο κρέας. Απάντησα, νομίζω, με βάση την προγενέστερη ερώτηση, αλλά αυτή η, βοηθή, ας το πούμε έτσι, η τεχνική, δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζουν τις ε, βασικές προδιαγραφές διατροφικής ασφάλειας δηλαδή ως προς τους ελέγχους υγείας και υγιεινής ή της ευημερία των ζώων και της υγείας των ανθρώπων δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ε, ελληματική προσέγγιση. Σε ορισμένα σφαγεία ε, πουλερικών και κουνελιών επειδή οι εθνικές αρχές πρέπει να εγκρίνουν την κάθε επιχείρηση, την κάθε μονάδα, σφαγής πουλερικών και κουνελιών. Επειδή θα πρέπει να γίνει λοιπόν αυτή η ξεχωριστή επιθεώρηση, αυτό θέτει προβλήματα για ορισμένα κρατημέλη που επέλεξαν αυτή τη λύση. Δηλαδή, όταν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εξαγωγές προς τρίτες χώρες, διότι πολλές τρίτες χώρες δεν αναγνωρίζουν αυτές τις προδιαγραφές θέλουν να υπάρχουν συνεχείς επιθεωρήσεις από ε, δημόσιους φορείς και αν υπάρχουν ιδιωτικές αρχές, ιδιαίτερα επιθεωρήσεις, ε, ως προς επιθεωρήσεις post-mortem, δεν θέλουν οι τρίτες χώρες να εισαγάγουν τα, τα πουλερικά αυτά ή τα κουνέλια. Κάτι το οποίο ε, θέτει επιπρόσθετες δυσκολίες στα κράτη-μέλη. Ως προς το τέταρτο ερώτημα, Ξέρετε ότι τον Νοέμβριο του 2009 το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τον εξυγχρονισμό επιθεωρήσεων ante-mortem και post-mortem στα ασφαγεία. Αυτό προς όλα τα ζώα, δηλαδή και τα μεγάλα ζώα και τα πουλερικά και κουνέλια. Υποβάλαμε ένα ερώτημα στην ΕΦΣΑ στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων για να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες του παρόντος πλαισίου και πώς μπορούμε να το αλλάξουμε και αναμένουμε απαντήσεις ε, μέχρι τα μέσα του 2011 ή μέσα του 2012 γιατί θα πρέπει να προσαρμοστούμε στην παρούσα κατάσταση καθότι όλοι οι κανόνες επιθεώρησης στα σφαγεία ορίστηκαν είτε πριν είτε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή δεκαετίες 50 το πολύ 60, με ασθένειες που δεν υφίστανται πλέον στα κρατη Εδώ αναφέρομαι στη φυματίωση των βοηδών που έχει εξαφανιστεί από, τα, από όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από δύο, όπου υπάρχουν ε, επιπτώσεις καθόλου αμελητές, αλλά έχει εξαφανιστεί από όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Άρα η ε, ανείχνευση αυτής της φυματίωσης είναι κάτι το περιττό πλέον. Η Εύσα θα μας πει κατά πόσο χρειάζεται ακόμα αυτή, αυτός ο ειδικό έλεγχος και η δεύτερη σειρά μέτρων αφορά την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και στις 18 Μαΐου του 2010 έγινε μία διάσκεψη όλων των αρχών επιθεώρησης και με, τα, και με τις τρίτες χώρες και στις 25 Οκτωβρίου θα γίνει μία νέα συνάντηση. Θα καλέσουμε και την Επιτροπή σας κυρία Πρόεδρε, να συμμετάσχετε σε αυτή τη διάσκεψη ή συνάντηση και να λάβετε το λόγο αν το επιθυμείτε. Αυτά, κυρία Πρόεδρε, αυτές είναι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των συναδέλφων σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διευθύντα. Ο κύριος Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την απάντηση που δώσατε στην επερώτηση η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία όλοι λάβαμε, <clears throat> είναι πράγματι καλή, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που βρίσκουμε εδώ στην Ευρώπη και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε κιόλα ότι αυτή η αλλαγή παραδείγματος την οποία επιφέρει ο νέος κανονισμός για την υγιεινή των τροφίμων όφιλε να γίνει και ότι αυτό πήγε καλά. Πρόκειται λοιπόν για πραγματική επιτυχία. Βέβαια εμείς θέσαμε την επερώτηση διότι ακριβώς αυτό που είπε μόλις τώρα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν φοβόμασταν και εμείς. Και γιατί θέλουμε λίγο να επισημάνουμε τον κίνδυνο αυτό. Είναι βέβαια αλήθεια ότι η οικονομική κρίση πλήττει όλους τους τομείς το ότι χρειάζεται εξοικονομήσεις παντού. Αλλά οι χώρες μέλη μέχρι τώρα και χωρίς οικονομική κρίση έκαναν σημαντικές εξοικονομήσεις στον τομέα αυτό. Δεν περίμεναν δηλαδή για να κάνουν εξοικονομήσεις να έρθει η οικονομική κρίση. Τώρα να τα φορτώνουν όλα στην οικονομική κρίση δεν με βρίσκει, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Γιατί για αυτή την ιστορία των ελέγχων την έχουμε παρακολουθήσει εδώ και καιρό στις χώρες μέλη, πάντοτε κάνει εξοικονομήσει σε αυτό τον τομέα. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου αμελούνται πλέον οι επιχειρήσεις, ή μάλλον οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις. Τώρα ας αφήσουμε λίγο τον τομέα του κρέατος. Μια επιχείρηση η οποία ελέγχεται μία φορά μόνο μέσα σε τρία χρόνια, τότε ας το ξεχάσουμε και αυτό τον έλεγχο, γιατί δεν υπάρχει απολύτως καμία επισκόπηση τη υγιεινή ε, στην πραγματικότητα σε αυτή την επιχείρηση. Άρα εδώ χρειάζεται να προβάλλουμε ένσταση, να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν, ότι οφείλει να υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις τους στις χώρες μέλη. Και αυτή βέβαια η μείωση του προσωπικού στις επιθεωρήσεις του κρέατος, επιθεωρήσεις του κρέατος που είναι απαραίτητες, να συνεχίζεται τώρα αυτή η μείωση του προσωπικού, μου φαίνεται και αυτή λάθος. Γι' αυτό η ε, ερώτησή μας. Γνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα και με το κρέας λαγών και πουλερικών και ορισμένων άλλων ζώων. Εγώ ίδιος έχω εργαστεί σε επιχείρηση παλαιότερα όπου η σχετική έλεγχη υπόκειταν στην κρίση του ίδιου του επιχειρηματία. Και γνωρίζω ότι πολλές επιχειρήσεις λένε την Κομισιόν ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε τους ελέγχους. Δεν μπορεί να είναι σωστό αυτό. Οι άνθρωποι που προσλαμβάνονται και εργάζονται στις επιχειρήσεις αυτές και αυτοί κοστίζουν χρήματα. Εάν τώρα τα χρήματα αυτά είναι λιγότερα, αν είναι φθηνότερη η λύση αυτή δηλαδή, το αμφισβητώ. Μπορούμε να κάνουμε άλλες συζητήσει για να δούμε πώ μπορεί να εξορθολογιστεί η εργασία αυτή. Οι περιφερειακές διοικήσεις καμιά φορά ας σημειωθεί φορτώνουν στις επιχειρήσεις με την ευκαιρία των ελέγχων και άλλα κοστολόγια τα οποία δεν εντάσσονται στην πραγματικότητα εκεί. Εκεί ίσω πρέπει να ξανασκεφτούμε τι μπορεί να γίνει. Αυτό ίσω είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσει στο μέλλον η Κομισιόν. Τώρα, μπορώ να φανταστώ όντω να δημιουργηθούν ιδιωτικοί φορεί οι οποίοι να προβούν στι επιθεωρήσει αυτέ, αλλά ω εξωτερικές, εξωτερικοί φορεί. γιατί αυτό είναι σημαντικό. Για τη βελτίωση των επιθεωρήσεων κρέατος νομίζω ότι η Κομισιόν κινείται στο σωστό δρόμο. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται ακόμα τώρα χρονολογούνται από πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εξέταση που γίνεται ακόμα τώρα δεν επιτρέπει να διαπιστωθεί η καλή υγεία του ζώου. Τώρα πια έχουμε διαφορετικές νόσους των ζώων, έχουμε διαφορετικά πράγματα που πρέπει να εξετάζονται. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας έτσι ώστε και να εξασφαλιστεί η υγεία του καταναλωτή, αλλά και να αντιμετωπιστούν και οι επιταγές της καθημερινής πραγματικότητας και βέβαια να διασφαλίζεται η σωστή εξέταση της υγείας των ζώων. Αυτά νομίζω θα είναι σημαντικό καθήκον και νομίζω επίσης θα επανέλθω τους απασχολουμένους της επιχείρησης. Εάν υπάρχουν προβλήματα εξαγωγών από τρίτες χώρες, θα ζητήσω εγώ από τις τρίτες χώρες να δραστηριοποιηθούν. Συνολικά λοιπόν θεωρώ ότι είναι εξαιρετική η ανακοίνωση της Κομισιόν με ικανοποιεί και το αποτέλεσμά της. Ας μην υποχωρήσουμε όμως τις πιέσεις των χωρών μελών που για λόγους κόστους ζητούν μειώσεις. Να ζητήσουμε από τις χώρες μέλη να τα αποκριθούν στα καθήκοντά τους να διεξαγάγουν πραγματικούς ελέγχους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την σκοπιά τη δική μου τουλάχιστον αυτό είναι το βασικό από τη σκοπιά του Ευρωβουλευτού δηλαδή. Ευχαριστώ Λίντα Μακάβαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις που έδωσε και για την δέσμευση που ανέλαβε ότι θα φροντίσει δηλαδή οι επιθωρήσεις της υγιεινής του κρέατος να είναι ε, θέμα προτεραιότητας και σε περίοδους κρίσεως το χρονοδιάγραμμα τώρα για τις νέες προτάσεις σας. Γιατί η πρόταση αυτή έχει μια ιστορία. Ξέρουμε ότι το 2004 οι χώρες μέλη, το Συμβούλιο δηλαδή, ήθελαν να παρατείνουν το καθεστώς επιθεώρησης των επιχειρήσεων και πέραν από το κρέας κουνελιών και ε, ορνήθων και στο βόλιο κρέας. Και ξέρω ότι ορισμένες χώρες μέλη πίεζαν πάλι για να αλλάξει το καθεστώς στις νέες προτάσεις και να ε, καταργηθούν οι ανεξάρτητες επιθεωρήσεις. Εγώ θέλω να μάθω, τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει προτάσεις με ορίζοντα 2011 και ξέρω ότι ε, εξελίσσεται η σκέψη αυτή της ε, Κομισιόν. Τι σκοπεύετε να κάνει έχοντας και υπόψη και τις εκθέσεις του FVO. Δεν θέλουμε, όπως είπε και ο Σνέλχαρτ, να φορτώσουμε και άλλο κόστος της επιχείρησης. Αυτά που μας είπατε όμως για προβλήματα με τις τρίτες χώρε και αυτά παίζουν ένα ρόλο εδώ. Εάν έχουμε τρίτε χώρε που λένε ότι δεν θέλουν να εισαγάγουν κρέατα από εμά γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στου εσωτερικού εσωτερικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις που κάνουν οι επιχειρήσεις, τότε αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να αλλάξει το σύστημα για το κόκκινο λεγόμενο κρέας. Δεν βοηθάει καθόλου λοιπόν οικονομικά την υπόθεση της Ένωσης εάν για λόγους οι οποίοι δεν είναι και γερά θεμελιωμένες και αλλιώς αλλάξουμε το σύστημα μπορεί να διευκρινίσει την θέση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι βέβαια το Κοινοβούλιο το 2004 δεν δέχθηκε την αλλαγή και δεν δέχθηκε να ξεφύγουμε από το καθεστώς των ανεξάρτητων επιθεωρήσεων. Άλλωστε γνωρίζουμε τι συμβαίνει όταν αποδυναμώνονται οι έλεγχοι της υγιεινής του κρέατος. Ξέρουμε τι συμβαίνει εν τέλει. Οι δε εξοικονομήσεις αυτές είναι πολύ μικρές σε σύγκριση εν τέλει με το τελικό αποτέλεσμα το οποίο είναι βαρύτατο για την υγεία των καταναλωτών. Πού, λοιπόν, προς τα πού σκέφτεται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς βλέπουν αυτό το θέμα με τις τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ Λίντα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τη δήλωσή τη. Ε, χάρηκα πολύ με κάποια από τα πράγματα που άκουσα. Συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους ότι το πραγματικό πρόβλημα εδώ είναι να διατηρήσουμε τα υψηλά πρότυπα κατά την επιθεώρηση των κρεάτων ε, στα σφαγεία. Και παρά τις αντιρρήσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, δεν ε, γίνεται πια η επιθεώρηση του λευκού κρέατος από ανεξάρτητους επιθεωρητές. Πιστεύω ότι, αυτό, ότι τώρα θα πρέπει να καλύψουμε και τον, το κόκκινο κρέας και να επιτρέψουμε στους στα σφαγεία να ορίζουν δικούς τους επιθεωρητές διότι θα υπάρχει έλλειψη διαφάνειας λόγω της έλλειψης ανεξαρτησίας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει αυτό. Μπορεί να αμφισβητηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος και όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση, κάποια από τα στοιχεία που είδα εγώ από διάφορους ε, φορείς που με έχουν πιέσει για το θέμα αυτό, διότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για το θέμα αυτό, ακόμα και σε αυτή την πρώιμη φάση της συζήτησης. Εάν ε, πρόκειτο να ε, αναθέσουμε στα σφαγεία την ευθύνη για να επιλέγουν εκείνοι τους επιθεωρητές τους, αντί να ε, έχουμε ανεξάρτητους επιθεωρητές και εάν εισάγουμε ελέγχους για να διασφαλίσουμε τα ίδια υψηλά πρότυπα, τότε ούτως ή άλλως το κόστος ε, θα είναι το ίδιο με, τους, ε, με το κόστος των ανεξάρτητων ε, επιθεωρητών. Δεν πρόκειται λοιπόν για πιο φθηνή επιλογή αν θέλουμε να διατηρήσουμε την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τα πρότυπα του κρέατος και των τροφίμων. Η ανεξαρτησία των επιθεωρητών διασφαλίζει τη δημόσια υγεία και διατηρούμε έτσι τα υψηλά πρότυπα πρότυπα. Στην Ουαλία, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, έχουν επιστήσει την προσοχή μου στα αποτελέσματα της τροποποίησης των κανόνων στο Ηνωμένο Βασίλειο του 2006 και η Κομισιόν παραπέμπει σε δικά της στοιχεία, τα οποία έχει συλλέξει από το Γραφείο ε, Τροφίμων και Εκτινιατρικών Θεμάτων. Και θα ήθελα να ξέρω τι θα γίνει με τα στοιχεία που ήδη έχουν παρουσιαστεί. Χαίρομαι που η Κομισιόν είπε ότι δεν προτείνονται τροποποίησεις αυτή τη στιγμή, παρότι εξετάζονται τα θέματα αυτά. Χαίρομαι που μου επιβεβαιώνει η Επιτροπή ότι, ε, ότι θέλει σύστημα ανεξάρτητων επιθεωρητών και ότι σίγουρα δεν θέλουν να μειώσουν τα πρότυπα, διότι αυτό είναι κάτι που ανησυχεί γενικά την Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο εδώ και αρκετό καιρό. Δεν θα ήθελα λοιπόν να κινηθούμε προς ένα σύστημα με πιο χαλαρούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Η κυρία Κλάση, Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω από αυτό που είπε η συνάδελφός μου προηγουμένως, ότι δεν πρέπει δηλαδή να αποδυναμώσουμε τις προδιαγραφές. Δεν μπορεί να είναι αυτή η πρόθεσή μας. Οι προδιαγραφές, τα πρότυπα, πρέπει να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο. Μιλούμε ιδιαίτερα για το κρέας και αυτό μας απασχολεί πολύ. Βέβαια, όταν μιλούμε τώρα εδώ για κρατικούς ή θεσμικούς ή ανεξάρτητους ελέγχους, ανεξάρτητος έλεγχος δεν σημαίνει ότι είναι κακός ή ε, οποιοδήποτε άλλος έλεγχος δεν είναι απαραίτητο λιγότερο καλός από τον κρατικό ε, έλεγχο γιατί και αυτό ο έλεγχος δηλαδή που θα διεξάγει μια ανεξάρτητη αρχή πάλι ε, θα υπακούει στα όσα επιβάλλει ο νόμος. στην περιφέρειά μου υπάρχει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό σφαγείο, το οποίο πλήττεται τώρα διότι καλείται να ανταγωνίζεται με σφαγεία άλλων χωρών μελών με διαφορετικές τιμές. Μπορεί να μας πει λίγο η Κομισιόν πώς σχηματίζονται οι τιμές αυτές και πώς φτάνουμε σε ένα επίπεδο τιμών πλέον που να προστατεύει και τους ελέγχους αλλά και να εξασφαλίζει και ανταγωνισμό. και ανάμεσα σε περιφέρειες και ανάμεσα σε κράτη-μέλη. Ο κύριος Πουτλέαν θέλει να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Πράγματι, θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα σημεία τα οποία ίσως δεν επεξήγησα αρκετά καλά. Στο ερώτημα των τριών Ευρωβουλευτών υπάρχουν τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι η χρήση βοηθών του ιδιωτικού τομέα για να αντικαταστήσουν τους δημόσιους υπαλλήλους στις επιθεωρήσεις στα σφαγεία. Η βασική υπηρεσία αφορά καταρχήν τους ε, δημόσιους κτηνίατρους και τους βοηθούς τους μπορεί να έχουμε δύο ή τρεις και 15 κύριους κτηνίατρους και γύρω στους 15 βοηθούς. Δεν μπορούμε να απαλείψουμε τη θέση του επίσημου κτηνίατρου διότι εγγυάται την ανεξαρτησία της επιθεώρησης, ιδιαίτερα αντεμόρτεμ, ελέγχει και η χνηλατή της ενδεχόμενης ασθένειας όταν φτάνουν τα ζώα στα σφαγεία και την ε, ε, ε, ζωή των ζώων. Και βεβαίως καταστρέφει το σφάγιο αν πρέπει. Ως προς τους επιθεωρητές του ιδιωτικού τομέα αντικαθιστούν αυτός του δημοσίου αλλά πρόκειται για βοηθούς που δεν έχουν πτυχίο της κτηνιατρικής σχολής και μετά από την νομοθεσία μας όπως συγκρίθηκε το 2004 ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει όσο αφορά τους ε, ε, ελέγχους του ε, επωνομαζόμενου κόκκινου κρέατος, των βοηδών δηλαδή κυρίως. Άρα αν θα πρέπει να αλλάξουμε τη διαδικασία θα πρέπει να έρθουμε ενώπιον σας στα πλαίσια μία συναπόφαση. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει επί του παρόντος. Δεν το επιθυμούμε επί του παρόντος. Δηλαδή ε, αυτό αφορά τα πουλερικά και όχι το κόκκινο κρέας. Δεύτερον, ο εξυγχρονισμός της επιθεώρησης που γίνεται από τον επίσημο κτηνίατρο, ιδιαίτερα στα βοηδή δεν αφορά δηλαδή τους βοηθούς που χρησιμοποιούνται στα σφαγεία πουλερικών. Υπάρχουν ορισμένες δράσεις που δεν θα σας περιγράψω εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε βεβαίως αν θέλετε. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά ε, δράσεων έτσι ως προς την ψηλάφιση των ζωτικών οργάνων του, του σηκωτιού, σπλήνα, καρδιά και ούτω καθεξής για να δούμε κατά πόσο με την ψηλάφιση αυτή υπάρχει μόλυνση και έτσι γίνεται και η ανείχνευση ασθενειών. Αλλά εδώ μιλάμε και για ασθένειες που δεν υφίστανται πλέον ή όχι πολύ πλέον. Δηλαδή, εάν δεν έχει ε, στην κοπή της καρδιάς των μειών ή του σηκωτιού, εάν δεν έχει αποστηρωθεί καλά το μαχαίρι, τότε δεν είναι σωστή η διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε από την ΕΦΣΑ να αποτιμήσει την όλη διαδικασία, έτσι ώστε να συζητηθεί με τις επίσημες αρχές και με τον ιδιωτικό τομέα. Και εδώ περιλαμβάνουμε και τον, την οπτική γωνία του καταναλωτή για τον οποίο προορίζεται αυτό το κρέας για να δούμε ακριβώς τι θα κάνουμε στο μέλλον. Άρα κατά τα μέσα του 11 ή 12, μετά από μία σειρά διασκέψεων, όπου θα σας καλέσαμε, θα σας καλέσουμε, θα καλέσουμε την Επιτροπή σας, θα αποφανθούμε για όλα αυτά τα θέματα, αλλά δεν θα γίνει αμέσως αυτό, θα γίνει μεσοπρόθεσμα. Θα ήθελα να απαντήσω ιδιαίτερα στις ερωτήσεις που υπέβαλε ε, ο κάθε βουλευτής. Ο κύριος Σνέλχαρτ μίλησε για έλεγχο κάθε τρία χρόνια. Όχι, στα σφαγεία γίνεται καθημερινός έλεγχος. Ο τριετής έλεγχος αφορά τις επιχειρήσεις που δεν είναι σφαγεία και όπου τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι υπάρχει ένας κίνδυνος ίσονος σημασίας ως προς το κόστος. Δεν θέλουμε να απαρνηθούμε τις κύριες επιθεωρήσεις εξαιτίας του κόστους, αλλά θέλουμε να βρούμε μια σωστή εξισορρόπηση μεταξύ του κόστους και της, του φόρτου των επιχειρήσεων, διότι έχουμε πολλές ΜΜΕ που έρχονται και μας προβάλλουν παράπονα ότι έχουν πολύ μεγάλο ε, φόρτο, οικονομικό δηλαδή. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε, να εξορροπήσουμε την κατάσταση έτσι ώστε να συμφιλιώσουμε την ανεξάρτητη επιθεώρηση, αυστηρή δηλαδή, που δίνει όλες τις εγγύσεις στον καταναλωτή και βεβαίως και τις εισφορές που θα πρέπει να καταβάλουν οι ΜΜΕ στον γενικό κρατικό προϋπολογισμό είτε στις υπηρεσίες επιθεώρησης. Ως προς τα ερωτήματα των κλάσμακ έβαν σε σχέση με τις τρίτες χώρες, σας είπα ότι αντιμετωπίσαμε προβλήματα με τις εξαγωγές πουλερικών, ιδιαίτερα προς, ε, ως από χώρε που χρησιμοποίησαν ε, οι βοηθούς που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και οι τρίτες χώρες δεν δέχτηκαν το κρέας που ήταν ε, απότοκο αυτών των ελέγχων με βάση το Κόντεξ Αλιμεντάριους που πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να ε, δεχτούν και δέχονται, πρόκειται για 160 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο που δέχονται αυτό το κώδικο, αλλά δεν αφορά το κόκκινο κρέας, δηλαδή κυρίως του, το βόιο και το μοσχαρίσιο καθώς και το πρόβιο. Η κυρία Κλάς ρώτησε τον, να της πούμε πώς υπολογίζονται αυτές οι εισφορές. Υπάρχει ο κανονισμός 882 που ορίζει την καταβολή εισφορών από τις διάφορες επιχειρήσεις και αναφέρεται σε παλαιότερες οδηγίες που υπάρχουν από το 75 και εφεξής. Η βασική αρχή έχει ως εξής. Οι εισφορές επίσημων επιθεωρήσεων ορίζονται με βάση το χρόνο είτε στα σφαγεία, είτε στις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις, είτε στις εκμεταλλεύσεις ε, παραγωγής ε, και ε, μεταποίησης προϊόντων μέχρι και τα εστιατόρια, γιατί θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο, μισθός ενός κτηνιάτρου, ο οποίος διαφέρει έφνης, είναι πολύ διαφορετικός μεταξύ Φιλανδίας και Ρουμανίας. Και υπάρχει ένα κατόφλι και μία οροφή καθορισμού αυτών των εισφορών. Δυστυχώς η πείρα μας μας δείχνει ότι επειδή τα κράτη-μέλη υφίστανται πίεση από τα Υπουργεία Οικονομικών, δυστυχώς οι εισφορές αυτές καθορίζονται, είναι μάλλον πολύ χαμηλές και δεν καλύπτουν το πραγματικό κόστος της επίσημης επιθεώρησης. Ενώ ε, αυτό είναι ο στόχος τις νομοθεσίες να καταβληθούν οι εισφορές έτσι ώστε να καλυφθούν τα έξοδα των επίσημων επιθεωρήσεων, η ε, κτηνίατροι, η μετάβασή τους ε, στις εκμεταλλεύσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηρίων και ούτω καθεξής. Αλλά για οικονομικούς λόγους τα κράτη-μέλη δεν ορίζουν τις εισφορές σε τέτοιο επίπεδο έτσι ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές δαπάνες των ε, επίσημων υπηρεσιών επιθεώρησης. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μία κατάσταση που αποκλίνει ανάλογα με, το κράτης, με τα κράτη-μέλη, σε μία αποκλίνουσα κατάσταση. Το 2011 θα αναθεωρηθεί αυτή η νομοθεσία. Είναι πρόωρο να μιλήσω γι' αυτό, γιατί τώρα γίνεται μια μελέτη αντικτύπου για να μπορέσουμε να επιλέξουμε μεταξύ της πλήρους απορρίθμισης έως ε, του καθορισμού εισφοράς που είναι παρόμοια για όλες τις ε, δραστηριότητες στα 27 κράτη-μέλη, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την διαφοροποίηση των μισθών. Είναι πολύ πρόωρο να σας πω αυτή τη στιγμή ποια λύση θα γίνει αποδεκτή από την Κομισιόν. Αυτά τα ολίγα. Ο κύριος Σνέλχαρτ νομίζω ήθελε να υποβάλει ένα ερώτημα. Ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα μου φαίνεται σημαντικό να μας προσκαλέσετε στις συνδιασκέψεις αυτές είναι σημαντικό να συμμετάσχουμε από την αρχή στην διαβούλευση. Το δεύτερο, και το βλέπω και καθημερινά στην πρακτική μου δουλειά στην εκλογική μου περιφέρεια, αναφέρεται στα τέλη, στις εισφορές. Και δεν νομίζω ότι οι δημόσιες αρχές θεσπίζουν πολύ χαμηλά τέλη. Εγώ βλέπω από την ίδια επιχείρηση να εισπράττονται τέτοιες εισφορές με διαφορά 50% και 100%. Το εύρος αυτό των τελών ή των εισφορών που μπορεί να εισπράξει η δημόσια διοίκηση, είπατε στο μέλλον θα ανταλλάξετε αυτά τα πράγματα. Το εύρος λοιπόν, αυτό το άνοιγμα αυτό πρέπει να μειωθεί, ώστε να μην υπάρχει αυτή η στρέβλωση του ανταγωνισμού που σημειώνεται αυτή τη στιγμή και που είναι σημαντική. Αυτό θα σημαίνει ότι ο φορολογούμενος ίσως καλείται να συμβάλλει περισσότερο, αλλά μην λησμονούμε ότι είχαμε και προτάσεις όταν συζητεί ο κανονισμός, είχαμε πει δηλαδή τότε θα αυτό το ποσό συν πλην ένα περιθώριο. Τέλος πάντων, τώρα έχω και μία ερώτηση, γιατί με απασχολεί το θέμα αυτό στην βάση. Εάν μία διοικητική αρχή θεσπίσει πολύ χαμηλές εισφορές, αυτό θεωρεί ότι, το θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι πολύ χαμηλές. Ή πάλι εάν επιστραφούν κάποιες φορές οι οποίες ήταν πολύ υψηλές, θεωρείται αυτό έμεση επιδότηση ναι ή όχι. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαριστούν έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μην οδηγούνται σε οικονομικές δυσχέρειες και ενδεχομένως και σε ε, πτώχευση λόγω των εισφορών αυτών. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε να αναμένουμε την πρόταση της Κομισιόν που σίγουρα είναι πολύ σημαντική και σίγουρα θα λύσει τα προβλήματα αλλά ε, για την ώρα σημειώνονται όλο και, όλο και περισσότερα καινούργια προβλήματα. Κύριε Μπουντλέ, μια τελευταία σειρά απαντήσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι κάπως περίπλοκη η κατάσταση στη Γερμανία, κύριε Σνέλχαρτ. Αφήσαμε την ελευθερία στις χώρες μέλη να ορίζουν αυτές τις εισφορές, οι ίδιες οι χώρες μέλη. Υπάρχει βέβαια και ομοσπονδιακός χαρακτήρας της ε, Ομοσπονδιακής Γερμανίας, όπου κάθε ε, κρατήδιο και κάθε διοικητική περιφέρεια θεσπίζει δικές της εισφορές, ώστε υπάρχουν αποκλήσεις στη Γερμανία. Όντως, που καμιά φορά είναι 50% παραπάνω ή παρακάτω από άλλες. Και μάλιστα και όταν και η ίδια επιχείρηση έχει εγκαταστάσεις σε περισσότερα από ένα ομόσπονδα κρατήδια. Αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία συμβαίνουν βέβαια κατά αναλογία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπα προηγουμένως ότι είναι πολύ ανομοιογενής η κατάσταση. Είναι αληθές αυτό αλλά το βλέπετε και μέσα στα πλαίσια της ίδιας της χώρας ε, μέλους, όπως η Γερμανία ή η Ισπανία. Για την ώρα δεν έχουμε ε, διαδικασίες επί παραβιάση, επί παραβάση, συγγνώμη, κατά χώρων μελών. Έχουμε ωστόσο επιβάλει υποχρεώσεις αποτελέσματος, δηλαδή να γίνονται επαρκείς επιθεωρήσεις στα σφαγεία για να διασφαλίζεται ότι το κρέας είναι καθαρό και από υγιή ζώα. Και κάθε ε, κυβέρνηση καλείται μετά να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις είτε να χρησιμοποιήσει δηλαδή, τις φορές των επιχειρήσεων είτε να χρησιμοποιήσει πόρους από τον προϋπολογισμό είτε του Ομόσπονδου Κρατηδίου είτε της Περιφέρειας και ούτε καθεξής. Ακόμα δεν έχουμε μπει στην δημοσιονομική συζήτηση εφόσον ε, ε, εφόσον οι εισφορές θεωρηθούν πολύ χαμηλές. Όπως είπα, δεν έχουμε ακόμα γύρει διαδικασίες επί παραβάση. Και πάντως σίγουρα οι εισφορές για τους κτηνατικούς ελέγχους δεν είναι αυτές που μπορούν να οδηγήσουν σε πτώχευση των επιχειρήσεων, γιατί το κόστος τους είναι ένα ή δύο λεπτά του ευρώ ανά κιλό κρέας. ακόμα και για τις επιχειρήσεις με μεγάλο τονάζ κρέατος, και εκεί δεν είναι οι επιθορήσεις, οι έλεγχοι οι οποίοι θα οδηγήσουν ενδεχομένω μια τέτοια επιχείρηση στην πτώχευση. Ίσως για κάποιες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις να είναι κάπως ε, βαρύτερα τα βάρια αυτά, κάπως σημαντικότερα τα βάρια αυτά. Εμείς θεωρούμε ότι η επιθεώρηση πρέπει να είναι υψηλή ποιότητας. Είτε την πληρώνει η επιχείρηση, είτε την πληρώνει το κράτος. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι λίγη εδώ η συζήτηση του θέματος αυτού. Τώρα υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα σχετικά με την έκθεση για την διατήρηση της βιοπικιλότητας, γιατί η συγκέντριά μας δεν έχει καταφτάσει ακόμα. Βρίσκεται ακόμα στο αυτοκίνητο. Γνωρίζετε βέβαια ποιες είναι οι δυσκολίες της κυκλοφορίας. Υπάρχουν ορισμένοι σκιώδεις ηγητές παρόντες στην αίθουσα, αν συμφωνείτε, μπορούμε να αρχίσουμε την συζήτηση, διότι αν δεν αρχίσουμε σήμερα, φοβούμε ότι αύριο λόγω φόρτου εργασίας δεν θα προλάβουμε και έχουμε και να ψηφίσουμε ε, γνωμοδότηση στις 14 Ιουλίου. Πρόκειται για έκθεση που δεν έχει νομοθετικό περιεχόμενο, που είναι όμως ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Ε, συμφωνείτε να προχωρήσουμε με τον τρόπο αυτό. Θα προτείνω λοιπόν στους σκιώδης ηγητέ όσοι εξ, εξ, αυτών το επιθυμούν να ζητήσουν να λάβουν το λόγο και στο μεταξύ θα έρθει και η εισηγητρία. Γιάν. Ευχαριστώ. Άρα μπορώ να μιλήσω ευθύς αμέσως. Ε, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που είναι απούσα όπως είπατε σχετικά με τα όσα έπραξε από την παρουσίαση του πρώτου σχεδίου της και μέχρι την κατάθεση των τροπολογιών της. Κατέθεσε πράγματι μερικές ε, σημαντικές τροπολογίες. Θα τις τα πω μετά βέβαια. Είναι σημαντικό ωστόσο και εγώ έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες, είναι σημαντικό πάντως να επιμείνουμε στους βασικούς στόχους. Πρώτα, ενίσχυση του ψηφίσματος. Εγώ πιστεύω ότι το κείμενο δεν ήταν αρκετά έντονο. Αυτή είναι η εξήγηση για ορισμένε από τι τροπολογίε μου. Επίση, να δώσω ένα πιο επίγοντα χαρακτήρα. Θεωρώ ότι η απώλεια βιοπικιλότητα δεν έχει συνειδητοποιηθεί ακόμα επαρκώ. ο κατεπήγον χαρακτήρας του θέματος. Επίσης, ήθελα να καυτηριάσω το, την έλλειψη πολιτικής βούλησης. Είδαμε και, στο, και, και στην παλαιότερη στρατηγική βιοπικιλότητας ότι με την εφαρμογή της δεν επιτύχαμε τους στόχους που είχαμε βάλει. Ένας από τους λόγους για αυτή την εξέλιξη είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης. Είναι δυνατόν να ανακοπεί η απώλεια βιοπικιλότητας εάν πράγματι το θέλουμε. Πρέπει να πηχεί όμως την πραγματική πολιτική βούληση. Τέταρτο, τέταρτος βασικός στόχος είναι ότι θέλω να τονίσω ότι χρειαζόμαστε καλύτερη εφαρμογή της σα ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας έχει ψηφιστεί και κυρωθεί, αλλά πρέπει να κάνουν περισσότερα οι χώρες μέλη για να την εφαρμόσουν. Τέλος, τελευταίο γενικό σχόλιο, ήθελα να τονίσω περισσότερο και τον οικονομικό, την οικονομική φύση της βιοποικιλότητας και μία από τις τροπολογίες μου αναφέρεται ειδικότερα στην πληρωμή υπηρεσιών οικοσυστήματος. Και ο τρόπος να ξεβρεθεί ιδιωτική χρηματοδότηση, γιατί ασφαλώς θα τη χρειαστούμε στο μέλλον. Εν τέλει, νομίζω επίσης ότι είναι σημαντικό να αναφερθούμε και στην συνδυάση που θα γίνει το φθινόπωρο στην Αγκόγια και να πούμε και σχετικά με το ψήφισμα, αλλά θα τα αφήσω για αργότερα αυτά. Έχω ακούσει έχω δει μάλλον ορισμένες καλές τροπολογίες της σχετικά με την Αγκόγια. Τέλος, έχω καταθέσει τις περισσότερες τροπολογίες μου μαζί με σοσιαλδημοκράτες συναδέλφους και από τους πράσινους και ανακαλύψαμε ότι μοιραζόμαστε πολλούς στόχους και ευχαριστώ τα πρόσωπα αυτά για την εξαίρετη συνεργασία. Ελπίζω να μπορέσουμε να επιτύχουμε να υπερψηφιστούν οι τροπολογίες αυτές, οι περισσότερες δηλαδή, από την Επιτροπή. Ο κύριος Αρσένης. Ε, Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών τονίζουμε την ανάγκη να εφαρμοστεί η αρχή της ε, προφύλαξης, όπως λέει το αφ 21, αρχή που είναι πια καθιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμο να μπει σε, όλους, σε όλα τα νομοθετικά κείμενα περί βιοπικιλότητας και να τονίσουμε ακόμα περισσότερο την ανάγκη να υπάρξει νομοθεσία ε, για βιοπικιλότητα όπως λέει και το 22 και όπως είπε ο κ. Γκερμπράντι να εξηγήσουμε για ποιο λόγο απέτυχαν οι πολιτικές μας αυτές μέχρι τώρα. Η έλλειψη δηλαδή πολιτική βούλησης, όπως είπε ο κ. Σκερβράντη, και η έλλειψη συνοχής των πολιτικών. Και αυτά τα λέμε στι τροπολογίε 15 και 34. Δεν χρειαζόμαστε μόνο νέου στόχους, αλλά χρειαζόμαστε νέου δεσμευτικούς στόχους, όπως λέει η τροπολογία 39, εν μέρη αποτύχαμε λόγω της έλλειψης δεσμευτικότητας των ε, στόχων μας. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε πλήρη εφαρμογή της οδηγίας Habitat και ένταξη των περιοχών Natura 2000, όπως λένε οι τροπολογίες 60 και 63. Άλλο σημαντικό για τις περιοχές Natura 2000 είναι ότι χρειάζεται να εξασφαλίσουμε την διασύνδεση των ε, περιοχών της Natura 2000, όπως λέμε στην τροπολογία 65, και επίσης, όπως λέει ο κ. Γκερμπράντι, να αναζητήσουμε τρόπους αύξησης της χρηματοδότησης. Η απόδοση των επενδύσεων στην βιοπικιλότητα θα είναι της τάξης του 200%. Και επομένως πόροι πρέπει να διατεθούν για την αποκατάσταση, όπως λέει και η σχετική τροπολογία, αλλά και η ε, βιώσιμη διαχείριση της Natura 2000, τροπολογία 140. θεωρούμε ότι και η, βιώσιμο, η βιώσιμη κατανάλωση έχει σχέση με τη βιοπικιλότητα και με την πολιτική για το 2020 και αυτό τα λέμε στην τροπολογία 138 γιατί τη Γεωργία τώρα έχουμε τέσσερα βασικά την ε, ε, τροπολογία 100 ε, ενίσχυση βιώσιμων πολιτικών στην Γεωργία για το ζωικό κεφάλαιο επίσης 107 τροπολογία και μαζί με την προστασία της βιοπικιλότητας απέναντι στους κινδύνους που προκαλούνται από την ευρεία χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Για τη βιοπικιλότητα λέμε για νομικά δεσμευτικά κριτήρια, τροπολογία 118, μιλούμε για κλιματική αλλαγή πάλι να ληφθούν μέτρα μετριασμού των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στη 129 τροπολογία. Επίσης για την ε, συνάντηση της Ναγκόγια, τροπολογία 180, και θέλουμε να περιληφθεί επίσης η βιοπικιλότητα και στους στόχους της χιλιετίας. Τροπολογία 189. Και υποστηρίζουμε επίση και αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο των μη κρατικών οργανώσεων. Προσθέτω επίσης ορισμένες τροπολογίες που συνυπέγραψα με άλλους συναδέλφους και θα τα συζητήσουμε μετά, αυτές τις μέρες δηλαδή στην ομάδα μας, για την διασύνδεση των προστατευμένων περιοχών χρειαζόμαστε ε, μια ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού υπέρ της ε, βιοπικιλότητας 122 το ίδιο για την διάβρωση εδαφών 135 και τελειώνοντας Έχουμε στις ιδέες της ταξινόμησης των οργανισμών αναλόγως με το αν είναι ωφέλιμα ή όχι για τον άνθρωπο. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι αρχή που πρέπει να υιοθετήσουμε. Και ταυτόχρονα το θέμα της μελέτης αντικτύπου που οδηγεί τελικά σε καθυστέρηση ανάληψη δράση σε ένα τέτοιο θέμα όπως ε, τον κινδύνο που απειλούν τη βιοποικιλότητα. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο, παρακαλώ. Φαίνεται πως όχι. Α, ο κύριος Πρόντι, με συγχωρείτε. Έχετε το λόγο. Το θέμα αυτό είναι μείζονος σημασίας και θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία των εδαφών για την στήριξη αυτών των ε, οικοσυστημάτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία, της, ε, το ρόλο της γης των εδαφών. Άρα θα πρέπει να έχουμε και ένα ειδικό νομοθετικό στοιχείο που να αφορά την διαχείριση των εδαφών και ίσως να διευκρινίσουμε κάπως καλύτερα τον ορισμό της βιοπικιλότητας, διότι θεωρούμε ως δεδομένο ότι πρόκειται για μία έννοια που γίνεται άμεσα κατανοητή. Όμως, για να ε, μπορέσουμε να μετρήσουμε τη βιοπικιλότητα και τις διάφορες εκφάνσεις της, χρειαζόμαστε μία συγκεκριμένη μεθοδολογία Άρα, ίσως θα μπορούσαμε να ε, προωθήσουμε περαιτέρω το ζήτημα από αυτή την έννοια της διευκρίνησης του ορισμού της βιοπικιλότητας και να δούμε ποιες είναι και οι συνέπειες των κλιματικών αλλαγών επί της βιοπικιλότητας. Ιδιαίτερα ε, υφίσταται το ε, θέμα του, της διάλυσης ανιδρυτών στο νερό και το στοιχείο της οξύτητας του ύδατος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και αυτό σχετίζεται και με την θέρμανση των ωκεανών. διότι έχει ε, μεγάλη σημασία αυτή η διαλυτότητα των ε, ανιδρυτών για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε την όλη κατάσταση ως προς το, την αλλαγή του, των κλιματικών συνθήκων. Θα πρέπει λοιπόν να διαθέσουμε περισσότερους πόρους για να φτάσουμε σε έναν καλύτερο ορισμό της βιοπικιλότητας γιατί χωρίς ε, μια τέτοια έρευνα δεν θα είμαστε ποτέ σε θέση να προωθήσουμε την ασφάλεια της βιοπικιλότητας και τη συντήρησή της. Σημεριζόμαστε την ε, άποψή σας, αλλά ξέρετε ότι η οδηγία για τα εδάφη έχει ε, για αρκετό χρονικό διάστημα. Θα ήθελα η Επιτροπή να απαντήσει, κυρία Κλόντια Λασαπάλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε επικροτούμε την έκθεση αυτή. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρη διότι βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι όσον αφορά την δημιουργία νέας πολιτικής για τη βιοπικιλότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μόλις υιοθέτησε την Άνοιξη νέο στόχο για μετά το 2010, για το 2020 δηλαδή, με νέο όραμα για το 2050. Ο νέος αυτός στόχος είναι πιο φιλόδοξος από αυτόν που έχουμε για το 2010, τον οποίο δυστυχώς ε, δεν καταφέραμε να πετύχουμε. Βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι δημιουργίας νέου πλαισίου, νέας πολιτικής που ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει αυτή τη φορά να πετύχουμε και να μην βρεθούμε το 2020 να ε, αναγνωρίζουμε ότι αποτύχαμε και πάλι, το οποίο θα ήταν πολύ κακό για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρισκόμαστε και σε σταυροδρόμιο όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικής, επίκυνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής, της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, της ε, πολιτικής συνοχής. Είναι τρία σημαντικά οχήματα. Θα πρέπει να ε, εξεταστεί το το, το δυναμικό για την προστασία του περιβάλλοντος. Ε, νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες συνδέσεις ανάμεσα στην έκθεση αυτή και σε αυτή που έχει να κάνει με την ε, μεταρρύθμιση της κοινή πολιτικής. πολιτική. Ε, συμφωνούμε απόλυτα με τις παρατηρήσεις για την ανεπαρκή χρηματοδότηση με τις παρατηρήσεις που έγιναν για την έλλειψη πολιτικής βούλησης και ευαισθητοποίησης. Συμφωνούμε απόλυτα ότι δεν έχει αναγνωριστεί το επίγον του προβλήματος. Ε, συμφωνούμε ότι είναι υψής της σημασίας να διασφαλίζεται η ε, πλήρης εφαρμογή όχι μόνο της ε, νομοθεσίας αυτής, αλλά γενικά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που επηρεάζει την βιοποικιλότητα. Πιστεύουμε ότι η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, διότι η Επιτροπή αυτή τη στιγμή δουλεύει δύο πράγματα. Την διαμόρφωση νέας ε, πολιτικής βιοπικιλότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που ελπίζουμε να ε, υιοθετηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα μετά την Αγκόγια και παράλληλα εργαζόμαστε σε διεθνές επίπεδο ώστε στην Αγκόγια να έχουμε ένα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο για την ε, Σύμβαση για την ε, Βιοπικιλότητα ε, και για το πρωτόκολλο EBS. Και σε διεθνές επίπεδο δηλαδή εργαζόμαστε εντατικά, διαμορφώνουμε και τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοπικιλότητα. Γι' αυτό επικροτούμε το ψήφισμα που ετοιμάζει το Κοινοβούλιο για την Αγκόγια. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε απόλυτα με τα όσα υπόθηκαν από αρκετούς ευρωβουλευτές. ότι είναι λυπηρό εάν δεν έχουμε οδηγία για το έδαφος, δεδομένου ότι ένας από τέσσερις ε, ζωντανούς οργανισμούς ζουν στο έδαφος, δεν θα πετύχουμε τους στόχους βιοποικιλότητας για το 2020. Άλλο σημαντικό κενό στην πολιτική είναι ε, τα επιθετικά είδη, τα οποία δεν ρυθμίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ε, βρισκόμαστε πίσω σε σχέση με τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία ή τις Ηνωμένε Πολιτείε. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε με τα άλλα θεσμικά όργανα, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και γι' αυτό επικροτούμε την έκθεση αυτή και επικροτούμε και τις πολλές τροπολογίες, 194 οι οποίες υποβλήθηκαν, που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον της Επιτροπής σας για το θέμα αυτό. Και αυτό είναι κάτι που επικροτούμε. Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο. Φαίνεται πως όχι. Λίγη συνεδρίαση και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Διότι δεν υπάρχουν άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη και η εισηγητριά μας δεν έφτασε εγκαίρως. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.